Good evening, colleagues. Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Σας παρακαλώ όλους να καθίσετε. Για να αρχίσουμε εγκαίρως, είναι πάρα πολύ αυστηρό το χρονοδιάγραμμα και θα πρέπει και να το τηρήσουμε. Καθίστε παρακαλώ και συζητήσεις εκτός της αιθούσης. για να μπορέσουμε να ακούσουμε ήσυχα τον Επίτροπο τον υποψήφιο και πρωταθέντα. Καλώς ορίσατε όλοι στη δημόσια αυτή ακρόαση. Εξ ονόματος της Επιτροπής μας θέλω να ε, καλωσορίσω τον κύριο Μίμητσα ε, που έχει προταθεί ως Επίτροπος για τη Διεθνή Συνεργασία και την Ανάπτυξη. Όπως γνωρίζετε το Κοινοβούλιο προετοιμάζει ε, την εκλογή της Νέας Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 118 και το παράρτημα 16 του κανονισμού μας αξιολογώντας όλους τους ε, ταθέντες επιτρόπους βάσει της γενικών ε, προσόντων, την ευρωπαϊκή προσήλωση και προσωπική τους ανεξαρτησία. Επίσης, εκτιμά το Κοινοβούλιο και αξιολογεί την κατανόησή τους και τη γνώση τους για το χαρτοφυλάκιο, καθώς επίσης και τις ε, επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Η παρούσα ακρόση έχει αυτό το σκοπό, είναι δημόσια και μεταδίδεται στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου και από το Europe by Satellite. Επίσης θα μαγνητοσκοπηθεί η ακρόαση και προσεχώς πολύ σύντομα θα είναι στη διάθεσή σας. Έχουμε διερμηνία σε 22 γλώσσες. Έχουμε πολύ αυστηρό χρόνο, αλλά σας παρακαλώ να μιλάτε με κανονική ταχύτητα. Μην προσπαθείτε να μιλήσετε πολύ γρήγορα, υπερβολικά γρήγορα, αλλιώ δεν θα σας προλαβαίνουν οι διερμηνείς. Και παρακαλείστε να κλείνετε το μικρόφωνο σας όταν τελειώνετε. Ο προτινόμενος επίτροπος έλαβε ένα γραπτό ερωτηματολόγιο έχει απαντήσει γραπτός, έχετε λάβει όλοι τις γραπτές απαντήσεις και διατίθενται επίσης ε, και συνέθουσα. Θα σας εξηγήσω λίγο τη διαδικασία. Πρώτα, ο, ο προτινόμενος επίτροπος θα κάνει την εισαγωγική του δήλωση που δεν θα υπερβεί τα 15 λεπτά. Η βασική ε, ακρόαση συνίσταται σε 45 ερωτήσεις από τους βουλευτές. Στο πρώτο γύρο θα ακούσουμε ένα εκπρόσωπο από κάθε μία από τις πολιτικές ομάδες. Οι ερωτήσεις αυτές θα είναι ενός λεπτού, όχι παραπάνω, και ο οριστής επίτροπος θα έχει 1,5 λεπτό για να απαντήσει. Μετά από κάθε ερώτηση μπορεί ο ερωτών να κάνει μια σύντομη συμπληρωματική μόνο για 30 δευτερόλεπτα και ο, ο, οριστή επίτροπο έχει ένα λεπτό για να απαντήσει. Όλες οι υπόλοιπε ερωτήσει θα είναι του ενό λεπτού και δύο λεπτά η απάντηση. Παρακαλώ να τηρήσουμε πάρα πολύ αυστηρά το χρόνο μα διότι δεν έχουμε ε, πολύ χρόνο. Θα έχουμε και δύο ερωτήσει από άλλε προσκληθήσεις επιτροπές, που είναι η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Επιτροπή ε, διεθνού Εμπορίου. Μετά τους συντονιστές θα λάβουν το λόγο και μετά ε, θα ακολουθήσουν οι ομιλητές των πολιτικών ομάδων. Αυτά είναι τα διαδικαστικά. Ελπίζω να πάει καλά η ακρόαση και με την ησυχία μας και ήσυχα να αφήσουμε τον κύριο Μίμητσα να μιλήσει. Έχετε το λόγο παρακαλώ για 15 λεπτά.